Ένας και θα δημοσιευτούν επίσης Θα ήθελα να σας ενημερώσω πως μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου συνυπέγραψα 18 νομοθήματα τα οποία εγκρίθηκαν με την τακτική νομοθετική διαδικασία. Όλα αυτά θα δημοσιευτούν στα πρακτικά αυτής συνεδρίασης. Περνάμε τώρα τις εργασίες αυτής της ε, συνόδου.